Και τώρα θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφων. Θα ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφων που δεν ε, μπόρεσαν να, να υποβληθούν χτες. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφων ως προς τη σημερινή ψηφοφορία. Το Πρώτο θέμα είναι πρόταση ψηφίσματος για την ε, κατάσταση στην ε, Μεσόγειο και την ανάγκη μιας ε, σφαιρικής προσέγγισης στο θέμα της μετανάστευσης. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Λούκε για ένα λεπτό. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Τζιλ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Φεράρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε προβλήματα σήμερα τα οποία έχουν να κάνουν με την, με την μετανάστευση στην ε, Μεσοή. Θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική αντιμετώπιση για να βρεθεί μια τέτοια λύση για το φαινόμενο. Έχουμε κάποιου φιλόδοξου στόχου που θα πρέπει να αντιστοιχούν σε κάποιο είδου δράσει για να καλυφθεί η να Θα πρέπει να δούμε ποια, ποια είναι η νόμιμη προσέγγιση και να σταματήσει η εκμετάλλευση και θα πρέπει να μην ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να ισχύει το κοινωνικό δίκαιο, ιδίω όσον αφορά τον οργανισμό του Δουβλίνου. Να εξεταστούν τα αιτήματα και θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και θα πρέπει να δούμε πώ θα καλυφθεί με κάποιου πόρου το άσυλο και η μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό στην Ιταλία γίνονται κάποιες έρευνες όσον αφορά τα συστήματα υποδοχής και τα σχετικά σκάνδαλα. Και αυτό θα πρέπει να ε, συνοδευτεί από τον έλεγχο της διαπλογής μεταξύ πολιτικών και των κυκλωμάτων διακίνησης. Θα πρέπει να γίνει επομένω μια εις συζήτηση και να δούμε πώς διαμορφώσουμε πολιτική για τη μετανάστευση και γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ του ψηφίσματος. Uh, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σούλτσε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η κατάσταση των προσφύγων στη Μεσόγειο γίνεται, επιδενώνεται συνεχώς. Ο πόλεμος του Ισλαμικού κράτους και η ευαίσθητη ε, κατάσταση στην ε, Αφρική, στη Βόρεια Αφρική οθεί όλο και περισσότερο, ε, περισσότερους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει βεβαίω να του βοηθήσουμε αυτού που θέλουν να μεταβούν στην Ευρώπη και όσοι βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη. Όλε οι χώρε θα πρέπει να αλληλοϊποστηριχθούν. Έτσι όπω το, βλέπει, ε, το προβλέπει η Συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 8. Βεβαίω θα πρέπει τα μεταναστευτικά ρεύματα να κατανεμηθούν σωστά. Αλλιώ επιβαρύνονται υπερβολικά ορισμένα κράτη. Καλό την Επιτροπή να το λάβει υπόψη, ε, κατά την χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής και να λάβει τα αναγκαία προς αυτό μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τζουφρίντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος γιατί πρόκειται για ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό βήμα ούτως ώστε να προσέξουμε περισσότερο αυτό το θέμα, αυτό το, το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης να σταματήσει η, υποκρισία, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι κατεπήγον, το αντιμετωπίζουμε σαν ρουτίνα, πρόκειται για μια αντίφαση και άρα δεν θα πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να μην αφήνουμε για αύριο ότι πρέπει να γίνει σήμερα και επομένως θα έχουν πολλά ακόμα να κάνουμε και ευθύ αμέσω θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η, η πολιτική στο μέλλον γιατί για το Μάρι νόστον δεν θα πρέπει θα να καταβληθεί να πέσουν στο κενό. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει, θα πρέπει και η Frontex να επιληθεί της ε, Σικελίας ε, εκεί όπου καταλήγουν πάρα πολλέ μεταστευτικές ροές. Βρίσκουν συνέχεια ε, ναι, ναι, θα πρέπει να βρεθούν διάβλοι για νόμιμη μετανάστευση και θα πρέπει να συνοηθούμε και με τις χώρες προέλευσης και να αποφύγουμε νέες ο κύριος Σεμπαστία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος γιατί ζούμε με άκρος δραματικό τρόπο τι συμβαίνει με τους μετανάστες. Εγώ προέρχομαι από την ε, Βαλένθια και ε, στο κόμμα στο οποίο εκπροσωπώ υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες από τη Θέουτα και την Μελίγια όπου βιώνουν καθημερινά αυτό το δράμα. Ε, θα πρέπει να δοθεί, ε, να σταθεί η παγκόσμια προσοχή στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ε, το ψήφισμα αυτό επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης ευθύνης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των χωρών προέλευσης, γιατί υπάρχει ανάγκη να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας συνεργασία. Γιατί μόνο μια πολιτική συνεργασία η οποία ε, υποστηρίζει τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ε, ζωής τους, μόνο μια πολιτική η οποία βελτιώνει ε, την κατάσταση στις χώρες αυτές θα μετριάσει τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Αρνουτού. Πρόεδρε, τη συνάδελφοι, όπως και το Εθνικό Μέτωπο, καταψήφισα το ψήφισμα που δεν αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή τελικά να ελέγξει τα 40.000 χιλιόμετρα ακτών και τα 9.000 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων των 28 κρατών μελών. Ακόμη και αν είχε την αρμοδιότητα. Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι. Από τη θέσπιση των συμφωνιών Σέγγεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε σε ό,τι αποπειράθηκε να υλοποιήσει τα εξωτερικά τη σύνορα. Ω εκ τούτου, κατακλυζόμαστε από παράνομους μετανάστε, οι οποίοι διαχέονται προ άλλα κράτη-μέλη στη συνέχεια και κυρίω στη Γαλλία. Κάθε εβδομάδα, περίπου χίλιοι μετανάστε διαβαίνουν τα γαλλο-ιταλικά σύνορα κοντά στην οικία που γεννήθηκα. Ήρθε ο καιρό να συναγάγουμε τα συμπεράσματά μα και να παγώσουμε αμέσω τη Συμφωνία Σέγγεν, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν πλέον τα σύνορά του. Is... Uh, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Παγκαζαουρτούντουα. She's Δεν παρευρίσκεται εδώ. επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ματέρα. She's not here either. Ούτε εκείνη παρευρίσκεται εδώ. Ας δοκιμάσουμε με κάποιον άλλον. Η κυρία Μλίνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ε, υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό για τη μεταναστευτική πολιτική, γιατί μια σφαιριστική προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης είναι ο μοναδικός ορθός δρόμος για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν σχέση με το θέμα της μετανάστευσης. Οι μεταναστευτικέ ροές είναι ένα διορθωτικό πρόβλημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και η πολιτική ασύλου έχουν ε, μεγάλη επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και η κατάσταση στη Μεσόγειο μας το αποδεικνύει κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν επιτακτικά να χαράξουμε μια νέα στρατηγική για την νόμιμη μετανάστευση. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας συστήσω την πρόταση της Αυστριακής Κυβέρνησης για την ε, κατανομή των μεταναστευτικών ροών βάσει μιας αρχής η οποία δράζεται στην αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Τόματσικ. Δεν βρίσκεται εδώ. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, τώρα είναι κάτι που όλοι δεχόμαστε ότι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη μετανάστε πρέπει να συντονιστούμε για πολλέ πλευρέ του προβλήματο. Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να προειδοποιήσουμε, πώ μπορούμε να κάνουμε μια συνόηση με τι χώρε αυτέ, τι χώρε προέλευση. Και θα πρέπει επομένω να γίνει ό,τι είναι δυνατόν να σωθούν κάποιε ζωέ. Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το τόσο επικίνδυνο ταξίδι και να σταματήσει η εκμετάλλευσή τους από τους εγκληματίες. Να βρούμε κάποιο είδους νόμιμους διάβλους για να φτάσουν στην Ευρώπη και να δούμε πώς μπορούμε να τους ε, εντάξουμε σε κάποιο είδους υποδοχή και στο σύστημα του ασύλου. Αυτό και είπαμε ότι αυτό το ε, ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε δεν είναι μια πλήρης απάντηση στο πρόβλημα. Είναι όμως ένα μικρό χρήσιμο βήμα. Δεν μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο, το ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με κάποια ε, μέτρα, κάποια μέτρα που θα έχουν προτεραιότητα και θα πρέπει επίσης να μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική που ήδη έχουμε χαράξει. Γι' αυτό και εμείς ψήφισαμε το ε, κείμενο. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ντεχόφσκι. Ε, κύριε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με το θέμα. Τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια απόφαση για τις μεταναστευτικές ροές. Το Συμβούλιο μετά από λίγο δημιούργησε την ομάδα εργασία για την Μεσόγειο όπου ε, το οποίο ακολουθήθηκε με ανακοινώσει της Κομισιόν. Θέλω να πω ότι η προσέγγιση μας είναι πολύπλοκη για ένα σύνθετο πρόβλημα όπου είναι δύσκολο όλοι να συμφωνήσουμε με όλα. Για το νέο έτος η ευχή μου είναι να επιδιώξουμε εξέβρεση λύσης όπου εμείς εδώ τα δημοκρατικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και όταν εμείς οι δημοκρατές δεν μιλήσουμε για την μετανάστευση θα αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο για τους λαϊκιστές. Κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει κανέναν. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Μωρέτη. Ευχαριστώ, βέβαια. αγαπητοί συνάδελφοι. Με ικανοποίηση μου να εκφράσω για αυτό που ψήφισαμε χτε. Θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική για την μετανάστευση, για να την υπάρχει ένα παράδεκτο. Κάθε μέρα αυτό είναι πιο βασικό. Κάθε φορά που έχουμε την τραγωδία στη θάλασσα χρειάζεται σφαιρική αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη. Και όλα τα κρατημέλη θα πρέπει συλλογικά να αναλάβουν την ευθύνη για αυτά τα θλιβερά συμβάντα. Αυτό θέλει δέσμευση, θέλει αλληλεγγύη, θέλει συγκεκριμένες αποφασιστικές κινήσεις και πρώτα πρώτα να παρεμβαίνουμε όχι στα αποτελέσματα αλλά στις ε, αιτίες, κάποιες απαντήσεις ούτω ώστε να έχουμε διάβλους νόμιμης μετανάστευσης και έτσι να αναπτύξουμε στρατηγική συνεργασία με τις τρίτες χώρες. το, το η Μεσόγειος έχει γίνει νεκροταφείο, γίνεται κάτι σαν ε, ομαδικό τάφος. Οπότε χρειάζονται επιγόντω, αποφάσεις αλλά και συνειδητοποίηση για όλες τις ε, χώρες. Ε, το ότι δεν πρέπει να διαχειρίζονται την κατάσταση μόνο οι χώρες που συνορεύουν, που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Τώρα έκθεση Μαμπίγεν, Ο πρώτος ομιλητή. είναι ο κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποφασίσαμε να συναυθεί αυτή η συμφωνία σύνδεση με την Γεωργία και εγώ είμαι υπέρ αυτή τη αποφάσεω γιατί έτσι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την εθνική κυριαρχία αυτή τη ε, χώρα ε, όπω και άλλε χώρε για όλα όσα έγιναν όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι τώρα επιβάλλουμε στη Γεωργία μια ιδεολογία ομοφιλόφιλη, λέω Και στη Γεωργία έχουμε χιλιάδες κατοίκους που στην Τυφλίδα κατέβηκαν σε συλλαλητήριο, σε διαμαρτυρία κατά αυτής της καταστάσεως. Καλύτερα θα πρέπει κάθε χώρα να έχει τη δική του τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα προβλήματα το ΕΛΚ δεν μπορεί να δεχθεί μια ε, νοοτροπία που αρμόζει στους ακραίους σοσιαλιστάς. Και αυτό άλλωστε αντιβαίνει και στους ε, ιδρυτές, στην των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Ποσπίσιλ τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο βουλευτής από την Τσεχία, μετά από την κομμουνιστική περίοδο, με αυτή την τραγική εμπειρία με τη Σοβιετική Ένωση. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι σήμερα εγκρίναμε και υποστηρίξαμε τη Συμφωνία Σύνδεση με τη Γεωργία. Έτσι, ανοίξαμε και τον δρόμο σε μια πρώην σιβηρική χώρα να ζήσει δημοκρατικά. Θεωρώ ότι το σχετικό ψήφισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αδύρυτη ανάγκη η πολιτική μας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει ακριβώς τους πρώην δορυφόρους της Κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης έτσι ώστε να γίνουν κράτη όπου θα βασιλεύει το κράτος δικαίου και ευημερία. Υποστηρίξαμε πρόσφατα την Μολδαβία, σήμερα υποστηρίζουμε την Γεωργία. Ευελπιστώ ότι η συμφωνία αυτή θα τελεί εποφελία του λαού της Γεωργίας και του κράτους δικαίου. Ήταν ένα βήμα απαραίτητο και χαίρομαι πραγματικά που έχουμε πλέον πολιτική, μια πολιτική προς την ανατολική μας γειτονία. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Σντάνοκα, είναι η επόμενη μιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά. Διότι σπέρνουμε έτσι την διχόνοια και όχι την ενοποίηση της Υπήρου με τον Νότιο Κάφκασο. η διατύπωση του κειμένου φοβούμαι ότι είναι ταπεινωτική. Η πρόταση να δημιουργήσουμε μια ειδική σχέση γειτονία με την Γεωργία στρέφεται κατά της Αρμενίας και του Ζαριμπατζάν. Η Ουσιατία και η Απχαζία αναφέρονται ως κατεχόμενες περιοχές και η Ρωσία ως εισβολέας. Ενώ ξέρουμε ότι οι Γεωργιανοί ξεκίνησαν τις εχθροπραξίες. Θεωρώ ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κίνηση αυτή. Συνεπώς, οι δηλώσεις ότι στόχος μας είναι η ευημερία στην περιοχή θα έπρεπε να είναι μια πραγματική δήλωση υπέρ όλων των χωρών της περιοχής και όχι μόνο μερικών. Αλλιώς τα πράγματα είναι πολύ αμφισβητήσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα τη συμφωνία γιατί όπως υπόθηκε πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Ε, πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει τον κόσμο. Μπορεί κανείς να τη βελτιώσει με εμπορικές σχέσεις και με αμοιβαίες σχέσεις σεβασμού και με τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δημιουργούμε εναλλακτικέ λύσεις για την περιοχή και βοηθούμε την βελτίωση της κατάστασης του κόσμου συνολικά. Και υπό την έννοια αυτή, αυτό είναι ένα βήμα για περαιτέρω συμφωνίες, σύνθεσης ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις δικές μας ε, πολιτικές ε, αξίες προς άλλες περιοχές του κόσμου, αντί να τις απομονώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάρ. Ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε αυτή τη κρίση στην Ουκρανία για να μας τυφλώσει αντί φαινομένων ε, ρεμβασισμού. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η Ρωσία συνεχίζει την κατάληψη μιας ε, κυρίαρχης ε, χώρας. Δεν πρόκειται μόνο για δαυκία καιρότητα, πρόκειται για μια προσάρτηση Πρόκειται για μία σύγκρουση την οποία είδαμε και στο παρελθόν μεταξύ, στην πρώην Σοβιετική Ένωση μεταξύ ε, ευρωπαϊστών, φιλοευρωπαϊστών και σλαβόφιλων εκείνων που επιθυμούν μια αυταρχική κοινωνία και εκείνων που επιθυμούν μια φιλελεύθερη κοινωνία. Ε, βεβαίως ε, τόσο για τους, το λαό της Γεωργίας όσο και για το λαό της Ουκρανίας ε, θα πρέπει να πάρουν τη δική τους ε, απόφαση. Αλλά αν αποφασίσουν στην κατεύθυνση των φιλελεύθερων δυτικών αρχών θα πρέπει να τις στηρίξουμε και δεν θα πρέπει να συνενέσουμε στην άσκηση βίας. ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο θα οδηγήσει σε νεοαπικισμό και θα υποστηρίξει τους συμπεριαλιστές του ημικυκλίου. Οι συνέπειες τώρα τα Χριστούγεννα θα ήταν κάτι το γελίο αν δεν ήταν τόσο τραγικές γιατί στο βορτιωτικό κομμάτι τη Αγγλία ε, είναι η εκλογική περιφέρεια λέγεται Stockport και χιλιάδες ε, από του ψηφόρους τώρα δεν θα, δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν θέρμανση, θα πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσει για να τραφούν και ενώ εσείς παίρνετε εδώ πέρα χρήματα και τα δίνετε σε δικτάτορες και παίρνετε επομένως την μπουκιά από το στόμα των ψηφόρων μας και τα δίνετε στους ε, άπλιστους της Γεωργίας και το UKIP και εγώ προσωπικά καταψηφίσαμε. Γιατί δεν πιστεύουμε στον εμπερισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παίρνει χρήματα από του φτωχού να τα δίνει στου πλούσιου. Δεν πιστεύουμε ότι ο λαό, ο κόσμο του στόχου θα περάσει Χριστούγεννα δυστυχισμένα, γιατί θέλουν να περάσουν Χριστούγεννα ευημερία οι πλούσιοι τη Γεωργία. Next speaker, Sean Kelly. Sean Kelly. Υποστήριξα την πρόταση από ομάδα μου. Πιστεύω ότι αποτελεί επίτευγμα την ευτυχή συσύμπτωση της παρουσίας δύο πρόεδρων εδώ για να γίνουν μάρτυρες αυτής της απόφασης του Δημοκρατικού Σώματος. Η πλειοψηφία υπερψήφισε θεμητή διαφωνία της μειοψηφίας. Και η Γεωργία ήρθε η ώρα να εκφράσει τις δημοκρατικές κρατικές της φιλοδοξίες και εδώ πρέπει να την υποστηρίξουμε. Πρέπει να τους δώσουμε χώρο εδώ στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό καταδηλώνει την βούλησή μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι λαοί θα ζουν ελεύθεροι και ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν ελεύθερες αποφάσεις σε όλον τον κόσμο. Είναι μια καλή μέρα για τη Γεωργία και μια καλή μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Και τώρα περνούμε σε μια άλλη έκθεση, σύσταση του κ. Αντρέη Μάμεκιν για την Συμφωνία Σύνδεση με τη Γεωργία. Ο κ. Πασπίσιλ έγινε ο πρώτος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, ήδη εξέφρασα την απόψή μου προηγουμένως. Να πω όμως ξανά ότι καλό είναι η συμφωνία να μην περιέχει μόνο οικονομικούς όρους αλλά να έχει στο κείμενο πέρα από τα τελωνία και το κράτος δικαίου στη Γεωργία την ενίσχυση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και πολλά άλλα. Είμαι πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη στην Τσεχία και γνωρίζω πολύ καλά ότι η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μόνο των οικονομικών θεμάτων αφορά και άλλα ζητήματα όπως ε, την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας, του κράτους δικαίου. Αυτά πρέπει να φροντίσει μια δημοκρατική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο κ. Κόμπερν. Ψήφισα κατά τη συμφωνία με τη Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομεί μια αυτοκρατορία, να κατέβεται στα χωράφια της Ρωσίας, όπως έδειξε η κρίση στην Ουκρανία. Δεν έφτανε αυτό. Τώρα μπλεκόμαστε και στην Γεωργία με αυτή την Συμφωνία Σύνδεσης. Η Γεωργία μέχρι και το 2008 ήταν σε πολύ μη κατάσταση με τη Ρωσία. Το UKIP πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά φασαρία στην περιοχή Η Ρωσία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση μαζί με το Ρούβλι και νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου σοφό να προκαλέσουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Πούτιν, ο οποίο παρά τι οικονομικέ δυσκολίε έχει περισσότερε μοιραρχίε τεθωρακισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία. Η Βερόνι Άστον, ένα επικίνδυνο ερασιτέχνη, ο πρώην Υπουργό μα ε, Εξωτερικών, πρόσφατα μίλησε για το φάσμα του πολέμου στην Ευρώπη. Εγώ θυμίζω ότι δεν θέλουμε το 1914 να ξανασυμβεί το 2014 στο πλαίσιο της οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη και ανόητη κίνηση να προκαλέσουμε τη ρωσική αρκούδα. Αγαπητοί τα πρακτικά της συνεδρίασης πρόκειται να υποβληθούν ε, διόντως για έγκριση στην επομένη